να προσθέτω βασίλειο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γεωούραβα για όλες τις απαντήσεις σας στα διάφορα μπλοκ ερωτήσεων. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Έχετε τώρα άλλα πέντε λεπτά και παρακαλώ να κρατήσετε το χρόνο των πέντε λεπτών maximum γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Έχετε λοιπόν αυτά τα τελευταία πέντε λεπτά για την τελική σας παρέμβαση έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδροι των Επιτροπών. Είμαι αρκετά κουρασμένη μετά από τρεις ώρες συζήτησης, αλλά θέλω να πω παρόλα αυτά ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τα ερωτήματά σας και να έχω τη δυνατότητα να σας δώσω την δική μου άποψη για τα θέματα αυτά. Σας είπα ότι είμαι πολιτικός κάποιες από τις απαντήσεις μου μπορεί να μην, να μην θεωρήσετε ότι είναι τόσο εξαντλητικές όσο θα περιμένατε από ένα τεχνοκράτη. Εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης, είμαι πολιτικός, αλλά προσπάθησα να σας δώσω τις απόψεις μου σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν το χαρτοφυλάκιο το οποίο, ε, για το οποίο υποψήφια της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ισότητας των φύλων. Νιώθω κάποια σύγχυση τώρα στο τέλος της ακρόασης και ξέχασα να βγάλω και το έγγραφο για την τελική μου παρέμβαση. Είμαι σίγουρη ότι θα ξεχάσω κάτι από αυτά τα οποία θέλω να πω. Κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό όμως και το οποίο δεν θέλω να ξεχάσω είναι το γεγονός ότι εάν μου δώσετε την ευκαιρία αυτή να είμαι η Επίτροπος για αυτά τα σημαντικά ζητήματα του χαρτοφυλακίου μου, και που οι δράσεις του επηρεάζουν όλο τον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαι ανοιχτή σε περαιτέρω συζητήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από κοινού και θα χαρώ πάρα πολύ αν μπορέσω να συνεργαστώ με όλους σας και ελπίζω ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και για την θετική ατμόσφαιρα, το θετικό κλίμα που δεν περίμενα κατά ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και η κυρία Πέρας Γκαρσία. Και τώρα θα πρέπει να κλείσουμε με τις παρεμβάσεις των προέδρων που έλαβαν μέρος σε αυτή την ε, ακρόαση με την ίδια σειρά που είχαν στην ε, ακρόαση αυτή. Ένα λεπτό κύριο Σφόμποντα. Ευχαριστώ κύριε θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου εκ μέρους της ε, Επιτροπής μας ότι έχουμε ε, αρκετές απαντήσεις στις ερωτήσεις για να προχωρήσουμε στη φάση αξιολόγησης της διαδικασίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τη γνώμη σας για το ζήτημα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και τα ζητήματα προστασίας του καταναλωτή. Μία παρατήρηση μόνο οργανωτικού χαρακτήρα θα γίνει η συνεδρίαση αξιολόγησης στις 6 στην αίθουσα ASP 5G3 και καλό τα μέλη, του συντονιστές της Επιτροπής Τρομικών Υποθέσεων στις 6 στην αίθουσα αυτή. 5G3. Αυτά από πλευρά μου και ευχαριστώ. Κύριο Μωράη, εκ μέρου τη Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών για του συναδέλφου που επέζησαν αυτή την ε, ε, μακροσκελή και έκτακτη συνεδρίαση και ευχαριστώ την κυρία Γιώργοβα. Για όσους λοιπόν είναι εδώ παρόντες, καταγράφουμε τη στράτευσή σας, δέσμευσή σας για συνεργασία σοντινισμένη με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς στο θέμα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, για συνεργασία με τους Άντσεπ για την... Ε, προσφέρει των καταναλωτών και το συντονισμό και σημειώνουμε τις απαντήσεις σε σχέση με το ε, ένταλμα συλλήψεως των δημόσιο κατήγορο, τους ε, νόμους για την κατάργηση των διακρίσεων κτλ. Και εδώ ακριβώς έγινε το πρόβλημα ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ε, και ταυτόχρονα πολύ επίτροποι θα συνεργαστούν σε συναφεί τομεί. Αυτό είναι πρόβλημα όχι δικό σα, είναι πρόβλημα δικό μα. θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πάντω αξιολογούμε με προσοχή τις απαντήσει σα. Θα πρέπει να σα ευχαριστήσουμε για το θέμα των προσωπικών δεδομένων. σα ευχαριστώ ιδιαίτερω που τοποθετηθήκατε σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα αξιολογήσουν βεβαίω τις απαντήσεις σα δηλαδή ε, οι συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σα. Κυρία Γιώροβα, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε απόψε για τις τοποθετήσεις σας. Είπατε στην καταλεκτική παρατήρηση ότι είστε πολιτικός και εμείς πολιτικοί είμαι και ως, είμαστε και ως πολιτικοί. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε μεταξύ μας, αλλά συμφωνούμε με τις αρχές της δημοκρατίας, ελπίζω. Και γι' αυτό και εγώ θα συναντηθώ με τα μέλη της Επιτροπής μου, τα οποία θα αποφασίσουν εάν έλαβαν επαρκείς απαντήσεις στα ερωτήματά τους και κυρίως αναφορά τα θέματα των καταναλωτών. Υπήρξαν ερωτήματα που προέκυψαν στο τμήμα που αφορά τη δική μου ε, επιτροπή που όμως δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της επιτροπής μου, κυρίως μία περίπτωση. Ε, λόγω λοιπόν του περίπλοκου χαρακτήρα του θέματος αυτού μπορεί να χρειαστεί η απάντησή σας στη συνεργασία και των άλλων επιτροπών. Αλλά τώρα θα προχωρήσουμε με δημοκρατικό τρόπο για να αποφασίσουμε εάν τα μέλη έχουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε μια αξιολόγηση. Και για να κλείσω εξ ονόματος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, θέλω και εγώ να επαναλάβω ότι όλοι οι συναδελφοί μου σας ευχαριστούμε. Έχουμε καταγράψει τις ε, απαντήσεις σας. Θα έχετε καταλάβει ότι είναι μια επιτροπή η οποία έχει πολύ απαιτητικό χαρακτήρα και πάντα έχει σταθεί κατά τη διάρκεια της οδηγίας αυτής. Γνωρίζουμε ότι 52% των Ευρωπαίων πολιτών είναι γυναίκες και δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση δεύτερης κατηγορίας. Και γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα παίξουμε το ρόλο μας στην αξιολόγηση και έχουμε κάθε θέληση να υπάρξει μια καλή συνεργασία για το καλό όλων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. και κλείνει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας για τη συμμετοχή.